τις αντιρρήσεις. Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, η δολοφονία των τριών ακτιβιστών Κούρδων γυναικών Σακινέκα Καζίτσε Ντοάν και Λελά Σονεμέτσε στο Παρίσι την προηγούμενη εβδομάδα μας συγκλώνησε βαθιά όλους. Εξ ονόματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στου γονεί των θυμάτων με μια επιστολή εξέφρασα τα θερμά μα συλληπιτήρια. Οι γονεί της ε, κυρίας Ντογάν, οι αδελφοί και τα αδέρφια της ε, ζουν στο Στρασβούργο και βρίσκονται σήμερα εδώ σε εμά στην Ολομέλεια. Σας χαιρετίζω στην Ολομέλεια και εξ ονόματος του σώματος σας εκφράζω τα βαθιά μας συλληπιτήρια. Ο θάνατος της κυρίας Ντογάν και των άλλων θυμάτων δεν θα πρέπει να μείνει ατιμόρυτος. Es gibt Προφανώς υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη διερμηνία, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε να δείτε αν είναι πρόβλημα με την ισπανική διερμηνία ή όχι. Ο θάνατος της κυρίας ε, Ντοάν, της κυρίας ε, Κανζίτσια και δεν πρέπει να μείνει ατιμόρυτη υπόθεση. Χαιρετίζουμε το στένος των ε, γαλλικών αρχών να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να διευκρινιστούν αυτοί οι φόνοι και να προσταθούν στα δικαστήρια υπεύθυνοι Κυρίες και κύριοι, μέλη της οικογένειας Άν, ξέρω πόσο δύσκολο είναι για σας αυτό. Είσαστε γείτονές μας στο Στρασβούργο και θέλουμε να σας πούμε και να εκφράσουμε ότι συμμεριζόμαστε τη θλίψη σας, όλοι μας. Κυρίες και κύριοι, οι αρμόδιες Ιταλικές αρχές ε, μου γνωστοποίησαν ότι ο κύριος Ροζάριο Κροτσέτα από την 17η Δεκεμβρίου 2012 διορίστηκε ως πρόεδρος της περιοχής της Σικελίας και από την κυρία Φραντσέσκα Μπαρατσού αντικαθίσταται.